Eh, Καλημέρα σε όλους και μας συγχωρείτε για την μικρή καθυστέρηση. Θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε το χρόνο, το χαμένο χρόνο, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες ε, θα κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Καθίστε για να ξεκινήσουμε. Βάσει του άρθρου 192 παράγραφος 2 του κανονισμού στι συνεδρίες των συντονιστών και στους αρμόδιους που μπορούν να συζητήσουν τα θέματα ανάθεσης εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων καθορίστηκε το πρόγραμμα ετήσιων εργασιών της Επιτροπής μας. Ο πρόεδρος Μπούζεκ με την έγκριση του Γραφείου της Προεδρίας ε, του Κοινοβουλίου ε, πρότεινε να ξεκινήσει μια διάσκεψη του δικτύου Σακχάροφ που είναι το δίκτυο των ανθρώπων που έχουν βραβευθεί με το βραβείο Σαχάροφ και θα συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις 23 Νοεμβρίου από τις 11 και μετά. Χρειάστηκε λοιπόν να αλλάξουμε την ημερομηνία της συνεδρίας της Επιτροπής μας που έπρεπε να γίνει τότε. Επομένως, η συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εκείνης της εβδομάδας θα ξεκινήσει στις 22 Νοεμβρίου το πρωί, αντί για το απόγευμα όπως είχε προβλεφθεί, και θα ολοκληρωθεί στις 23 Νοεμβρίου στις 10.30 προκειμένου να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την αίθουσα για την διάσκεψη η οποία θα γίνει στην ίδια αίθουσα. Εξ ονόματος ε, του Προέδρου φυσικά είστε όλοι προσκεκλημένοι ε, και ζητούμε για την ενεργό συμμετοχή σας στην διάσκεψη αυτή. Θα σας διανεμηθεί και το πρόγραμμα σύντομα. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να έχετε έτοιμες τις κάρτε σας, από ό,τι βλέπω περισσότεροι είστε ήδη έτοιμοι. Ένα λεπτάκι να προετοιμαστούμε και θα ξεκινήσουμε εντό ολίγου. Καλώ. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτη ψηφοφορία, Πρόοδο που σημειώνει η εφαρμογή τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κεντρική Ασία. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 η οποία θα γίνει κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα και μόνο διευκρινιστικά να σας πω ότι το δεύτερο τμήμα αφορά τον όρο conditional. Δεύτερο τμήμα λοιπόν, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Conditional. Chiusa. Πέρασε της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι κατά, 30 υπέρ, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Περνάμε Στην τροπολογία 25 ως και με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, α... εγκρίνεται. 26, 27 και 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την ε, τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία; 29 κατά, 25 υπέρ, απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεν πέρασε, οπότε ψηφίζουμε την 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 41. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα αν δεν ε, σηκώνετε τα χέρια σας. Πέρασε της ψηφοφορίας 34 υπέρ 19 κατά είναι μεγάλη πλειοψηφία. Εγκρίνεται λοιπόν. 42-43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 25-31 εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά. Δεν είναι σαφές ε, το αποτέλεσμα της 50. Να ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 28-28. Πράγματι λοιπόν, δικαίως δεν ε, είχα καταλάβει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το τελευταίο γκολ στα πέναλτι. Το λύσαμε. Με μία ψήφο λοιπόν υπέρ εγκρίνεται η τροπολογία 50. 51 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 52 υπέρ. Συγγνώμη να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 51. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία η ψήφο σας την προσμετράμε και έχουμε και πάλι το πέναλτι της κυρίας Γιαννάκη 29-28. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα της 54. Άρχεται η ψηφοφορία για την 54. Τέσσερις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Αφηρημένοι είστε βλέπω. Λείπει μία ψήφος. Εντάξει. 29, 28 και μία της κυρίας Γιαννάκη 30. Γιαννάκου, συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50, 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63. Να ελέγξουμε την 62. Ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία για την 62. Πέρας της ψηφοφορίας. 28-29 και υπάρχει και η δεύτερη ψήφος κυρίας Γιαννάκου με δύο ψήφους διαφορά λοιπόν εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64. Δεν την ψηφίσουμε. 65 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα τη 68. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορία. 29 κατά, 28 υπέρ. Προστίθεται η ψήφο, η οποία από τούδε και στο εξή θα είναι ηλεκτρονική, γιατί περνάει η κάρτα. 29-29 όμω απορρίπτεται. Αυτή τη φορά όμω, παρά την προσθήκη τη ψήφου, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, συγγνώμη, ε, τροπολογία 71 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 78. Πέραση ψηφοφορίας. 30 ψήφοι κατά, 29 υπέρ. Απορρίπτεται. 79 γιατί δεν εγκρίθηκε 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα μία προφορική τροπολογία για την τροπολογία 96. Θα μας την παρουσιάσει κάποιος ή να τη διαβάσω εγώ. Ο κύριος Κυρίλοφ είναι παρόν. Θέλετε να μας πείτε την προφορική σας τροπολογία. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια προφορική τροπολογία για το ότι τελευταία έχουμε θετικά νέα για πιθανή συμφωνία με το Τουρκμενιστάν και το Αζερβαϊτζάν για ένα έργο αγωγού από την Κασπία. Οπότε η τροπολογία μου 11α τονίζει την ε, μεγάλη σημασία του έργου αυτού για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης και εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την στήριξή του για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα. Σημειώνει με ικανοποίηση την ετοιμότητα Τουρκμενιστάν ε, για να υπογράψει μια συμφωνία. E Πρόκειται για προσθήκη δηλαδή, ε, δεν τροποποιεί την ε, τροπολογία, να ακούσουμε όμως ε, την γνώμη της εισηγήτριας, η κυρία εισηγήτρια. Η πράσινη δεν είναι υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε την προφορική τροπολογία, επομένως δεν το ψηφίζουμε. Τροπολογία 97 συγγνώμη, 96 χωρίς την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Επομένω ψηφίζουμε την 105 με ηλεκτρονικό τρόπο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. 29 κατά, 30 υπέρ, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 109. Πέραση της ηλεκτρονικη ψηφοφοριας ψηφοφορίας. Πράγματι. 50-50 το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται λοιπόν 110 και 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά δεν είναι σαφές άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για την 118 πέραση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 25 κατά 34 υπέρ εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125. Ωραία. 125 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Υπάρχει μια προφορική τροπολογία που θέλει να παρουσιάσει η συγγήτρια. Παρακαλώ, κυρία Λίζα. <laughs> Η κυρία Γέγκερ, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν τη συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τονίζει πως οι συγκεκριμένες ε, παράγραφοι των ε, εξή χωρών ε, περιέχουν κάποια σημαντικά ζητήματα αλλά δεν έχουν στόχο να δώσουν μια πλήρη συνολική ανάλυση της κάθε χώρας. Bene. Καλώ. Πρόκειται για μια διευκρίνηση λοιπόν. Υπάρχουν ενστάσεις. Όχι. Δεν υπάρχει καμία ένσταση. Ωραία. Δεχόμαστε την προφορική τροπολογία προς ψήφιση λοιπόν ε, και ψηφίζουμε unblock την, ε, τις τροπολογίες και την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. με την προφορική τροπολογία που έγινε παραδεκτή και την έχουμε συμπεριλάβει στην ψηφοφορία. Ναι, με την ψηφική τρο... τροπολογία. ancora una decina di deputati. Ecco, adesso stiamo chiudendo. Bene. Sì, sì, no. Adesso... Ολοκληρώνεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία, μεγάλη πλειοψηφία, 50 υπέρ 9 κατά εγκρίνεται. 132. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 132. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν σας βλέπω να σκόνετε τα χέρια σας. Πέρασε τις ψηφοφορίες. 27 κατά, 29 υπέρ, εντάξει και διανατάσσεως χειρό, δεν θα καταλάβαινα. Πέρασε πάντως, 133 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 135 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 136 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται, 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 138-139 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Θέλετε επαλήθευση. 138 και 139 λοιπόν, άρχεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Ένας δεν έχει ψηφίσει, 29 υπέρ, 28 κατά και μία αποχή. Ωραία, εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ. Ζητώ συγγνώμη. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία για την 141. Πέρας ψηφοφορίας. 29-29 είναι συνέχεια το σκορ. Απορρίπτεται λοιπόν. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 Ελέγχουμε λοιπόν την 155. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 29-29 και πάλι. Απορρίπτεται λοιπόν. Ισοψηφία. 156 υπέρ. Κατά. Μπορεί να έχουμε την ίδια διαφορά, αλλά να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 156. Με έχετε βάλει σε μπελάδες σήμερα. Μισή-μισή πρέπει να προσέχω περισσότερο. Λείπουν τρεις βουλευτές, δεν έχουν ψηφίσει. Μπορεί να μην θέλουν να ψηφίσουν. Πέρασε ψηφοφορίας. 25 κατά 30 υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 162 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 169 να ελέγξουμε την 168. Ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ένας δεν έχει ψηφίσει, πέρασε της ψηφοφορίας. 26-29 εγκρίνεται με τρεις, αποχέ ε, με τρεις αποχές. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 170. Πέραση της ψηφοφορίας. 26-29. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 174. Θέλετε να κάνουμε παλήθευση για την 172. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 37-22 εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 σας παρακαλώ όμω, σηκώντε τα χέρια σας. 174 να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα ήθελα σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί χάνουμε χρόνο. Να ψηφίσω κι εγώ. 174 πέραση της ψηφοφορίας. 2632 εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 175. Αυτή τη φορά δεν φταίτε εσείς. Πέρας της 32 32-27 απορρίπτεται. Πάμε στην 176-77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180-81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183-84 θέλετε να ελέγξουμε την 182 ωραία ηλεκτρονική επανλήθευση για την 182 Τρει συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Δεν πειράζει. Πέραση τη ψηφοφορία. 25-29 εγκρίνεται. 183, 84, 85 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τις 183, 84 και 85. Πέραση ψηφοφορίας 24-35 εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές απο, εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, συγγνώμη, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 5. Πέραση τη ψηφοφορίας. 25-34 εγκρίνεται.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 αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα της 18. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 18. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 29 ψήφι κατά, 28 υπέρ, απορρίπτεται. Είναι τα δύο της γνωμοδότησης υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία για την ίντα 2. Chiusa la 24. Πέραση ψηφοφορία 24-35 εγκρίνεται. Είναι 3 υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Είναι 9 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Είναι 12 υπέρ κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Είναι τα 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. DV5 θέλετε να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την DV3. La... Πέραση της ψηφοφορίας για την DV3. 24 κατά 34 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ε, διακρίνω καλά το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για την 5. ΔΕΒΕ 5 Πέρασε της 35 «35-23 εγκρίνεται». Δεν ψηφίζουμε την 6 γιατί ε, την ροφά η συμβαστική τροπολογία 5, 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ΔΒ 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω να κάνουμε μια επαλήθευση μισό λεπτό διακοπή Ε, eh, Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή. Πρέπει να κάνουμε ένα reset ε, που θα χρειαστεί κάποια λεπτά. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μια ψηφοφορία ανατάσσεως χειρής, αλλά ήταν λίγο δύσκολο να δούμε το αποτέλεσμα. Ε, ψηφίζουμε την ΤΕΒΕ 12. Υπέρ λοιπόν για την ΤΕΒΕ 12.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 Ci sono delle Αποχές. Τέσσερις αποχές. Φαίνεται λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι 27 25 υπέρ. Ελπίζω να μην είχαμε κάνει λάθος ε, στην καταμέτρηση, γιατί με δύο ψήφους διαφορά, αν θέλετε να είμαστε πολύ αυστηροί και να περιμένουμε τον ηλεκτρονικό έλεγχο, μπορούμε να περάσουμε. Αν ε, δεν θέλετε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Δύο ε, ψήφοι είναι μικρή διαφορά. Δέβε 14, υπέρ. Βότι κοντράρι. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δέβε 15, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 17 όχι. Εδώ όμως τώρα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ψηφίσουμε το ψήφισμα ως τροποποιήθηκε. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, η τελική ψηφοφορία θα γίνει όταν θα έχει ε, επαναξεκινήσει η συσκευή κατά μέρους των ψήφων και θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση που και πάλι έχει η συγκίτρια την κυρία Κιλ Νίλσεν. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Τώρα λοιπόν που λειτουργεί η συσκευή μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 59 ψηφίσατε, 35 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ωραία. Ελέγχουμε την τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 43-15 απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 18 υπέρ, τη 17 θέλετε να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Νομίζω πως η 16 καταπίπτει. Η 17 όχι. Την 17 ψηφίζουμε, τη 16 δεν την ψηφίσαμε. Η τροπολογία 16 δεν ψηφίστηκε γιατί κατέπεσε. Εάν ε, έγινε λάθος στη μετάφραση, εγώ ούτως ή άλλως έθεσα προς τη 17. 43 κάτι. Η 17 απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. 21 υπέρ. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. ψηφοφορία. 35 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. Συγγνώμη, αλλά δεν είδα. Σωστά. Α, όχι. Είχα πει ότι εγκρίνεται. Δίκαιο είχα. Δίκαιο είχα. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφής η 5, άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιο δεν ψήφισε. Πέρασε ψηφοφορία. 31 ψήφι, 31 ψηφί υπέρ, 28 κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική ψήφο. Κάποιο ε, έχει βάζει την κάρτα του και δεν ψηφίζει. Πέρασε τη ψηφοφορία λοιπόν. 56 ψήφοι υπέρ, καμία αρνητική ψήφος και καμία εποχή εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την έκθεση για τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρικής Ασίας ε, που είχαμε αναβάλει. Ψηφίζουμε λοιπόν, επειδή είχαμε διακόψει προηγουμένως για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, είμαστε πάντα με λιγότερου ψηφίσαντε. Περιμένω ένα-δύο δευτερόλεπτα, αλλά αν ξεχνάτε να ψηφίσετε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα κλείσει η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. 49 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Δύο λεπτά διάλειμμα για να ε, ανασκουμποθούμε και συνεχίζουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ και μην ξεχάσετε τις κάρτες.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 Ωραία, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας παρακαλώ καθίστε. Είμαστε στο σημείο υπαριθμών 6 της ημερήσιας διάταξης, ε, δημοσιομελωμικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Γιάτεν Μάκη. Έχουμε 24 τροπολογίες οι οποίες παρουσιάστηκαν από τους συναδέλφους Μα ενδιαφέρει ο έλεγχο του προπολογισμού για τη χρηματοοικονομική υποστήριξη στο Αφγανιστάν και είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο χωρί περαιτέρω καθυστήρηση στην ε, συντάκτρια για να μα ενημερώσει για τα τη γνωμοδότησή τη και τι ε, τροπολογίε που κατατέθησαν. Παρακαλώ κυρία Γιατανμάκη. Thanks, Λοιπόν, η διεθνή κοινότητα είναι παρούσα στο Αφγανιστάν από το 2001 και δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί και υποσχεθεί στη χώρα, αλλά τα αποτελέσματα είναι περιχρά. Αλλά η κατάσταση ασφαλείας και ο πόλεμος βεβαίως είναι ένα σοβαρός λόγος για τη χαμηλή αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Με λύπη μου σημειώνω πως πολλοί αναπτυξιακοί δείκτες δεν δείχνουν ακόμα σοβαρή βελτίωση. Οι βασικές προκλήσεις με τη βοήθεια στο Αφγανιστάν είναι πως η βοήθεια δεν φτάνει πάντα τους δικαιούχους τους οποίους θα θέλαμε, δηλαδή τον αφγανικό λαό και η κοινωνία συχνά ασκούμε κριτική στους Αφγανούς για διαφθορά και δικαίως. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε πως και εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Είναι απολύτως αναγκαίο η Κομισιόν και η διεθνής κοινότητα να δώσει μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο στο κόστος των ενδιάμεσων. Εμείς ζητάμε ένα κεντρικό σύστημα πληρωμών και να αναλύσουμε επίση το κόστο και αντίκτυπο τη βοήθεια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω πω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν ε, επικαιροποιημένα και αξιόπιστα δεδομένα και έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της βοήθειας. Τέλος, θέλω να τονίσω πως είναι αναγκαίο η Κομισιόν να επιμείνει σε επαρκή πληροφορίε για τα αποτελέσματα και τη χρήση των κονδυλίων, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω πως εάν εισαχθεί τομεακή στήριξη του προπολογισμού στο Αφγανιστάν μπορεί να δοθεί μόνο σε διοίκηση η ικανότητα οικονομικής διαχείρισης της οποίας έχει κριθεί διαφανής θέλω να τονίσω πως ε, δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά εάν δεν υπάρξει κάποια αύξηση της ε, διοικητικής ικανότητας. Συνάδελφοι από διάφορες ομάδες κατέθεσαν συνολικά 24 τροπολογίες. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν πως υπάρχει ο τίτλος «Καταπολέμηση διαφθοράς και ανάγκη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας». Και εγώ κατέθεσα κάποιες τροπολογίες μαζί με τους σκιώδεις ε, εισηγητές Αρλάκη και Τισέτ και εδώ πέρα βασιζόμαστε λοιπόν στη βελτίωση, διαφάνεια και λογοδοσία καθώς και την ε, κατάργηση της καλλιέργειας οποίου. Θέλω και την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους κυρίους Λάτκη και Λίζεξ για την πολύ καλή συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαρίστω να δεχτώ σχόλια επί της γνωμοδότησης και των ανθρωπολογιών. Σας ευχαριστώ κύριε Γιατανμάκη. Κύριε Αρλάκη. Uh, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι η γνωμοδότηση αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν στον τομέα της χρηματοοικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να τονίσω ότι αυτή η γνωμοδότηση ε, περιέχει τη κοινή θέση διαφόρων ομάδων, το επιβεβαιώσαμε και για άλλη μια φορά συγκλίνουν οι απόψει σχετικά με την ανάλυση τη ανθρωπιστική βοήθεια προς το Αφγανιστάν. Αυτά δηλαδή ε, που ε, εμπεριείχε και ένα ψήφισμα που ψηφίσαμε πριν από ένα περίπου χρόνο εδώ στο Κοινοβούλιο. Τονίζεται όλο ιδιαίτερο στη γνωμοδότηση ότι υπάρχει ένα πελώριο πρόβλημα διαφθορα ε, και διασπάθηση κονδυλίων από, από πλευρά του Αφγανιστάν. Ε, δηλαδή ε, διασπάθηση των κονδυλίων που προέρχονται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά γενικότερα από την ε, διεθνή κοινότητα. Είναι μια συμβαστική λύση ε, στην οποία κατέληξε ήδη από πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής δυστυχώς ε, δεν έχει δοθεί καμία συνέχεια ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από το Συμβούλιο παρά την τραγωδία που βιώνει σήμερα το Αφγανιστάν. Ευελπιστώ λοιπόν ότι σύντομα θα έχει την ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει εκτενέστερα αυτό το θέμα. Μία αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Αφγανιστάν. Όλα τα προβλήματα, όλες οι αρνητικές εξελίξεις ε, θα ληφθούν δεόντως υπόψη, κυρίως ως προς τα ζητήματα ασφαλείας. Ευχαριστούμε κύριε Αρλάκη. Ο κύριος Λίζικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε εδώ μέσα πως η βοήθεια του Αφγανιστάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και από τρίτες χώρες είναι κάτι το οποίο βεβαίω πρέπει να συνεχιστεί για πολλά χρόνια γιατί έτσι είναι η κατάσταση του Αφγανιστάν και εμείς διεθνή κοινότητα έχουμε αναλάβει ένα μερίδιο ευθύνη για το μέλλον αυτής της χώρας. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω τα λόγια των συναδέλφων που ήδη ομίλησαν. Δηλαδή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιατεμάκη για την καλή συνεργασία είναι ένα καλό έγγραφο το έγγραφο το οποίο έχουμε. Οι μεγάλες πολιτικές ομάδες συμφωνούν με αυτή τη γνωμοδότηση. Οι βασικές τροπολογίες είναι κοινέ τροπολογίες, κάτι το οποίο είναι ένα σαφές μήνυμα για το ότι οι απόψεις μας συμπίπτουν. Θα ήθελα να τονίσω την τροπολογία 14 η οποία δηλώνει πως ε, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βοήθεια των κρατών μελών και η βοήθεια των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να συντονίζεται με άλλους δωρητές όπως η και η Ιαπωνία για να μην σπαταλάμε λεφτά να ξοδεύονται σωστά τα χρήματα. Ευχαριστούμε κύριε Λίζεκ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν έχει κάποια παρατήρηση η συγκήτρια. Συγγνώμη, δεν σας είδα. Παρακαλώ. Η κυρία Λέζινγκ. Δεν σας είχα στον κατάλογο ομιλητό. Ε, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως η ομάδα μου και εγώ ήμασταν εξ αρχής κατά του πολέμου στο Αφγανιστάν και το έχουμε πει πολλές φορές ε, στην Επιτροπή αυτή. Είναι πραγματικά άσχημο Ο πόλεμος αυτό συνδέεται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, τρομοκρατία. Αλλά αντιθέτως δεν έχουμε νικήσει έτσι τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τρομοκρατία. Η έκθεση τώρα βεβαίω είναι ισορροπημένη και σας ευχαριστώ. Έχω καταθέσει μόνο μια συμπληρωματική τροπολογία η οποία επαναλαμβάνει το αίτημά μας τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούνται μόνο για μη στρατιωτικά μέτρα. Δηλαδή να μην εκπαιδεύεται ο στρατιωτικός και αστυνομικός μηχανισμός. Και μια που αναφέρθηκα στον αστυνομικό μηχανισμό, συμφωνώ με τη λογική της κυρίας Γιατενμάκη, πρέπει να σκεφτούμε ποιο καθεστώς εδώ πέρα εξοπλίζουμε με μέσα καταστολής και αυτός ο αστυνομικός μηχανισμός στρέφεται κατά του πληθυσμού του Αφγανικού και ε, είναι πολύ πιο φοβερή αυτή η αστυνομία από πολλές άλλες. Ευχαριστούμε κυρία Λέζινγκ. Δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις τώρα. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο η συντάκτρια για να ολοκληρώσει. Όχι. Ωραία. Η μόνη ανακοίνωση λοιπόν που πρέπει να σας κάνω είναι ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ήταν η 29 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι και ψηφίζουμε στις 20 Οκτωβρίου. Καλώς, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας και θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 ε, με κεκλεισμένο των θυρών ε, συνεδρίαση για την εκλογή του Τετάρτου Αντιπροέδρου. Σας ευχαριστώ. Εσάβριον είναι το σπουδαία. Καλό βράδυ.